από την GUNGL τον διορισμό σε κοινοβουλευτικές επιτροπές θα περιέλθει στα σημερινά πρακτικά η πρόταση αυτή και αν δεν υποβληθούν περαιτέρω παρατηρήσεις μέχρι να εγκριθούν τα πρακτικά αυτά οι διορισμοί αυτοί θεωρούνται ότι εγκρίνονται.